Good afternoon, uh, um, συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Θα προσέξατε ότι σήμερα έχουμε κάποιους φιλοξενουμένους εδώ στο Προεδρείο. Έχουμε επίσης και την πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης για το επόμενο θέμα. Και επίσης έχουμε και κάποιους βουλευτές, συναδέλφους από τον Νίγερ για το επόμενο θέμα. Θα τα πούμε μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έχουμε επίσης και τον πρέσβη της χώρας. Οπότε πρώτα απ' όλα έχω κάποιες ε, ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα έγκριση της ημερής διάταξης. Ε, δεν υπάρχει ένσταση, εγκρίνεται και τώρα έχουμε μία σειρά ανακοινώσεων. Πρώτα πρώτα έχουμε, μόνο δεν θα έχουμε από και ισλανδικά και ελτικά την ερμηνεία και επίσης έχουμε γράψει προτάσεις των συντονιστών ε, διάταξη 2.05 να εγκρίνουμε πρώτα πρώτα όσον αφορά την ε, ανταπόκριση την απόκριση τέλο πάντων ε, το τι έγινε στις συνεδρίσεις της Τετάρτης του 5ου επίσης έχουμε τον ορισμό εισηγητών για τους Ισλαμοκράτες ο κύριος Μάμπηγινς για την πρόταση εικονισμού όσον αφορά τη θέση σε εμπορία και χρησιμοποίηση των προδρόμων εκρηκτικών επίσης για την συμφωνία καθεστώς Frontex ο κύριος Βαλέρο και ο Ζωράντεφ επίσης ε, για μια οδηγία η οποία θα θεσπίζει κανόνες για διευκόλυνση ε, χρηματοοικονομικών και πληροφοριών όσον αφορά την πρόληψη ε, ποινικών αδικημάτων. Επίση, ο κ. Γκουριάνο από το ΕΛΚ είναι ο για την ε, πρόταση της απόφασης του Συμβουλίου για κάποιο είδους κατάργηση θεωρήσεων διαβατηρίων. Επίσης για τις ε, γνωμοδοτήσεις. Ο κύριος Σντεχόφσκι του ε, ΕΛΚ, εισηγητής για την εφαρμογή των διδάξεων της συνθήκης όσον αφορά την αναβαθμισμένη ενισχυμένη συνεργασία. Ε, αυτό είναι έκθεση της της ΑΦΚΟ. Συμφωνείτε, μάλιστα. Οπότε τώρα, άλλες ανακοινώσεις όσον αφορά κάποιο είδου κατανάθεση και εφαρμοστικές πράξεις. Ζητώ την υπομονή σας για να δούμε αν χρειάζεται όλα αυτά να τα διαβάσουμε. Ναι, είστε βεβαίως. Καλώς. Θα είναι αυτό λίγο βαρετό, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό από ό,τι μου λένε, επιβάλλεται. Οπότε, λίγη υπομονή. Έχουμε τώρα αυτέ τι εφαρμοστικέ και κατανάθεση κατεξοδότηση πράξη 25 του 18 το Κοινοβούλιο έλαβε το σχέδιο εφαρμοστική απόφαση που θεσπίζει κάποια μέτρα για την ε, θέση εφαρμογή του συστηματο entry Entry-Exit System. Επίσης, ε, για Καλλιδονία, Πολυνησία, ε, κάποια σχετική απόφαση για διάφορες περιοχές τέτοιες. Επίσης, 25 Μαΐου έχουμε μια προθεσμία ε, εσωτερικής υποβολής ενστάσεων. Ε, οπότε αν κάποιος έχει κάποια ένσταση να το πει πριν τις 8 Ιουνίου στην Γραμματεία. Τώρα έχουμε για μια εφαρμοστική απόφαση όσον αφορά βιομητρική επαλήθευση και ταυτοποίηση για το σύστημα Entry Exit, EES. Ε, δεύτερον, εφαρμοστική απόφαση για κάποια μέτρα προσβασιμότητας των σχετικών δεδομένων του ΙΕΣ. E e ε, επίσης, σχέδιο αποφάσεως της Κομισιόν για ε, σβήσιμο, διαγραφή δεδομένων του ΙΕΣ. E Τέταρτον, για το ΙΕΣ πάλι συγκεκριμένες διατάξεις. Ε, πέμπτον, έχουμε εφαρμοστική απόφαση που θεσπίζει τις ε, προϋποθέσεις, τα προαπαιτούμενα της, ε, των επιδόσεων του ΙΕΣ και τελευταίο οι προδιαγραφές για το Μητρό Δεδομένων του ΙΕΣ πριν τις 8 Ιουνίου τις ενστάσεις σας παρακαλώ προς την γραμματεία μας. Επίσης, άλλες ανακοινώσεις, 31 Πέμπτου, σχέδιο εφαρμοστικού, εφαρμοστικής αποφάσεως, συγγνώμη, αφορά τους κανόνες λειτουργίας του πάνελ της Επιτροπής Επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 για το γραφείο για την υπηρεσία του Ευρωπαίου ε, Εισαγγελέως. Και εδώ έχουμε κάποια προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Επίσης, έχουμε στις 35 τις εφαρμοστικές αποφάσεις για την αξιολόγηση του 17 όσον αφορά το SIS, το Σύστημα Πληροφοριών Σέγγεν. Και αυτά διαβιβάστηκαν σε ένα newsletter σε όλους τους συναδέλφους τον Ιούνιο. Επίσης έχουμε κάποιες ε, συστάσεις όσον αφορά προβλήματα του συστήματος 16 ε, και 17 έγινε η αξιολόγηση για την εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν ε, για Πορτογαλία, Μάλτα, Στονή και Σουηδία. Ήδη είμαι κουρασμένο. Δεν ξέρω εσεί πώ θα πάτε. Σα ευχαριστώ για την υπομονή σα. Επαναλαμβάνω, επιβάλλετε αυτά να τα ε, διαβάζουμε εδώ. Τι να κάνουμε. Αυτά επιβάλλει η πειθαρχημένη μας οργάνωση. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 3. Και όπως είπα στην αρχή, με μεγάλη μου χαρά, θα σας παρουσιάσω τους ε, συναδέλφους που έχουν έρθει. Πρέπει να ευχαριστήσω πρώτα τη Λίντα Μάκαβαν, την πρόεδρο της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης που θα μας συνοδεύσει σε αυτή την ακρόαση, μια που η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, είναι αρμόδια για ένα σωρό θέματα που αφορούν τον Νίγηρα. Οπότε θα μας τα πει κατά την ακροασή. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Σαμινού Λάουλη που είναι βουλευτής από την χώρα αυτή. Και επίσης τον κύριο Αγκάλη. Και εσείς καλωσορίσατε ορίσατε αγαπητοί συνάδελφοι τα είπαμε στην χώρα σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία και για το ότι εξασφαλίσατε την ε, επιτυχία της αποστολής. Αλλά έχουμε και τον πρέσβη Ματέους Παύλα, τον οποίο και ευχαριστούμε που και αυτός συνέβαλε στην επιτυχία της δύσκολης αυτής αποστολής. Και πάλι ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η στιγμή για την Επιτροπή μας, διότι όπως και η Επιτροπή θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα για αυτές τις χώρες που περνάνε τόσο βαθιές αλλαγές και πρόσφατα επίσης είχαμε και στη Λιβύα μια ε, αποστολή όπου και εκεί ε, η δουλειά μας ήταν ε, παρόμοια σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Πάντως τα βασικά εκεί είναι η ανθρωπιστική βοήθεια και επίσης μια σφαιρική προσέγγιση στα ζητήματα. Ε, γι' αυτό ακριβώς και κάνουμε αυτή την ακρόαση από κοινού με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Οπότε, επίσης, θα πρέπει να καλωσορίσουμε έναν ειδικό του Οργανισμού Μετανάστευσης, τον κύριο Κεσάντα. Επίσης, την κυρία Αναμπέλ Ροϊ Γκράνιον, που υπηρετεί την ύπατη αρμοστία πρόσφυγης του ΙΕ, τον Ντένις Αβό που είναι διευθυντής του Ερυθρού Σταυρού ε, και την Σουμαίλα Εμπρέμ που είναι συντονίστρια για τα θέματα ιατρικής ε, σε σχέση με τον ε, Νίγηρα από πλευράς των γιατρών του κόσμου του Βελγίου. Όπως σας είπα, Πήγαμε 20 23 Μαΐου στην ε, Λιβύη και θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή περίληψη των πεπραγμένων και θα δώσω τη στην κυρία Λίντα Μάκαβαν για να σας τα πει για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Όντως είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται στα θέματα τα σχετικά με την ανάπτυξη και τη μετανάστευση οι ε, επιτροπές μας η ιδιαίτερη πολιτική έμφαση δίνεται αυτή την εποχή, ιδιαίτερα σε σχέση με την Ιταλία. Υπάρχει όμως όλο και περισσότερη χρηματοδότηση για τις πολιτικές, για τη μετανάστευση στις χώρες εταίρους και βέβαια όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική διάσταση και ειδικότερα την ε, μετανάστευση παίρνουν μεγαλύτερη και υψηλότερη προτεραιότητα. Είναι βέβαια πολύ σημαντικός εταίρος ο Νίγηρας στην ε, προσπάθεια αυτή. Θα ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας ασφαλώς. Ο τίτλος της ακρόασης είναι πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τον Νίγηρα. Ένας από τους καταλληλότερους τρόπους πιστεύω είναι η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός εταίρος ε, του Νίγηρα. Είχαμε πρόσφατα την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου στη συνεδρία στη συζήτηση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αύξηση πρότεινε την αύξηση κατά 90 εκατομμύρια ευρώ της διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας. Από 596 εκατομμύρια δηλαδή πάμε τώρα στα 686 εκατομμύρια ευρώ, μεγαλύτερο τμήμα των οποίων υποστηρίζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη των κοινωνικών πολιτικών από τις κυβερνήσεις. Ε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί από αυτούς που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για να μεταναστεύσουν ε, το πράττουν γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες. Το μεγαλύτερο λοιπόν τμήμα αυτής της βοήθειας θα πάει στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ένας άλλος τομέας όπου επενδύουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα καταπιστεύματα, 230 εκατομμύρια σε 11 διαφορετικά έργα στην, ε, στον Ήγυρα, επί παραδείγματι, και χωρίς να έχω επισκεφτεί τον Ήγυρα τον ίδιο, αλλά μόνο την ε, γειτονική Ουγγάντα, βλέπω ότι έχουμε να κάνουμε ένα σημαντικό έργο, μια προοπτική ανάπτυξη σε έργα, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινή ζωή του πολίτη. Και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα όταν πρόκειται για μετανάστε ε, βελτίωση όχι μόνο τη ζωή του μετανάστη του ίδιου, αλλά όλη τη κοινωνία στην οποία ζει, όλων των πολιτών. Βεβαίω το Κοινοβούλιο έχει ρόλο την, ε, ε, τον έλεγχο, την εποπτεία της χρήσης αυτών των καταπιστευμάτων και των κονδυλίων τους με την Ελισλάιν αρμόδια Χαίρομαι ιδιαίτερως που βλέπουμε εδώ μεταξύ μας και βουλευτές αφρικανικών χωρών. Την ίδια υποπτία δηλαδή πρέπει όπως και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκούν και οι Αφρικανοί ομολογοί μας. Στην κοινοβουλευτική συνέλευση της Αμπιτζάν κάναμε μια συνάντηση ε, με ταξί Ευρωβουλευτών και Αφρικανών ομολόγων μας και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ως πολιτικοί πώς θα διαχειριστούμε τα ζητήματα αυτά. Βεβαίω περιμένουμε να ακούσουμε από εσά τι θέσει σα ε, και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τι εξελίξει τη ε, χώρα σα και ποια θέματα βλέπετε ότι χρειάζονται περισσότερη συνεργασία. Εν τέλει, έχουμε να κάνουμε με μια πολύ σημαντική εβδομάδα για την αναπτυξιακή πολιτική, με τις ε, ημερίδες για την αναπτυξιακή πολιτική που οργανώνουμε σε μια μεγάλη διάσκεψη που θα ε, παρακολουθήσουν πολλοί άνθρωποι για να συζητήσουν τα θέματα της αναπτυξιακής πολιτικής. Την Τετάρτη προβλέπεται ένα ειδικό ε, θέμα συζήτησης για τους ε, γάμους ανήλικων παιδιών με εκπροσώπους και από τον Ιγύρα. Αυτό το οργανώνουμε εμείς. Χαίρομαι λοιπόν που σας βλέπω σήμερα εδώ. η κοινοβουλευτική αυτή, η διακοινοβουλευτική αυτή συνεργασία, συνεργασία με τους βουλευτές από τον Ήγηρα πιστεύω ότι θα έχει τις καλύτερες δυνατές, ε, την καλύτερη δυνατή απήχηση και αντίκτυπο. Ευχαριστώ πολύ Λίντα, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω αυτά που είπες για τη χρηματοδότηση. Θεματά μετανάστευση στοχεύουν αυτές οι, μετα... οι χρηματοδοτικές ροές, αλλά όπως είπαμε πρέπει να υπάρξει και μια αλλαγή προσέγγιση. Το είδαμε άλλωστε και στη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδας για τη Λιβύη. Και οι συνάδελφοι ζήτησαν μια σύντομη ε, επικαιροποίηση ενημέρωση για την αντιπροσωπεία που μετέβει στην Λιβύη με μεγάλη σημασία για την ε, Επιτροπή μας, για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ενημερώσω και μετά θα περάσουμε στο θέμα του Νίγηρα. Όπως είπα, είναι θέμα σχετικό, γιατί λάβαμε μέρος στην αποστολή αυτή για πρώτη φορά μετά το 2012 για να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις. μετά τις επισκέψεις τη κυρίας Μογκερίνη και τη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ στο να σα ενημερώσω λοιπόν τι συμβαίνει, τι συνέβη. Ε, στο κομμάτι της αντιπροσωπεία που επισκεφθήκαμε την Τρίπολη. Ενημερωθήκαμε για την κοινωνική πολιτική κατάσταση. Προφανώς αν δεν υπάρχει σταθερότητα κοινωνική πολιτική μέχρι τις εκλογές, πριν τις εκλογές τα πράγματα θα είναι πολύ σοβαρά και άρα μας ε, ενδιαφέρουν όχι μόνο τα θέματα τα προφανή που είναι η μετανάστευση και θα περάσω βέβαια και σε αυτά αμέσω, αλλά και το θέμα της σταθερότητα. σταθερότητας. Για τον Ήγηρα η μετανάστευση, η διαχείριση μετανάστευσης είναι ένα θέμα το οποίο ε, μας έχει απασχολήσει και στο θέμα της ε, Λιβύης. Συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό και τον ε, αναπληρωτή Πρωθυπουργό, τον Πρωθυπουργό Σιάλα, τον ε, Δήμαρχο Πτώργα. δήμαρχο μια πόλη 5.000 κατοίκων που ακόμη δεν έχουν μπορέσει να επιστρέψουν στι αιστείε του ύστερα από την αναγκαστική του φυγή ε, όταν του εκδίωξαν ε, τα μέλη τη διοίκηση τη Μισράτα. Το κέντρο κράτηση Τάρικαλ Σίκρα επίση επισκεφθήκαμε. Οι συνθήκε ήταν αποτρόπε, ήταν εφικτέ για μας. Φυσικά αυτό μπορούμε να το συστήσουμε και σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά έκρινα απαραίτητο να σας ενημερώσω για την επίσκεψη αυτή. Καλούμε την Λιβική κυβέρνηση να αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα για να κλείσουν τα κέντρα αυτά. Το επαναλάβαμε άλλωστε και στη συζήτηση επί τη ευκαιρία της εκθέσεως Παντζέρη την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Τίνιδα γιατί είχαμε πολλά άλλα γεγονότα, θα είμαι όμως ωστόσο τον πιο σύντομο για να περάσουμε στα θέματα του Νίγηρα. Στην Τίνιδα λοιπόν είχαμε ε, συζητήσει ε, συζητήσεις με εκπροσώπους των Εθνών για την ε, πρόταση του ειδικού εκπροσώπου Σαλάμ των Εθνών ε, μιλήσαμε με πολλές με κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη, δεν είναι και πολλές, με την Amnesty International, με τους ε, ιατρούς χωρίς σύνορα, για τη δράση τους σε στεριά και τη θάλασσα. Μιλήσαμε για την ανάγκη να ε, τεθεί ένα τέρμα στην πολιτική αστάθεια και αναταραχή και να τηρηθεί η προθεσμία για την διεξαγωγή εκλογών το 2018, που δεν είναι πιθανό να τηρηθεί. Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λιβύη, είναι πολλές οι αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων ομάδων, με θύματα αμάχους, με πολύ εμφανή κλιμάκωση της κατάστασης. Το επισημάναμε αυτό σε κάθε ε, συνάντησή μας με αξιωματούχους. Όπως είπε και η Λίντα, είναι πολλά τα προβλήματα, πολλές οι άνθρωποι που χάνονται. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες στο Νότο. Επίσης σε κάποιες περιοχές όπου ε, υπάρχει ακόμη δυνατότητα εξόρυξης πετρελαίου ε, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μιλήσαμε για την ε, πολύ σημαντική συγκέντρωση πυροβόλων όπλων που είναι μάλλον η υψηλότερη στον κόσμο, στις περιοχές Λιβύης και θα συνεχίσω πολύ γρήγορα για να πω ότι είχαμε επαφές και με την ακτοφυλακή. Πρέπει νομίζω να ε, πούμε ότι επαναλήφθη η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έργο της ακτοφυλακής που πρέπει να έχει πρώτη στο μέλημα την ασφάλεια και όχι μόνο τη φύλαξη των συνόρων. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης ε, των ε, ε, προσφύγων, των άνθρωπινων δικαιωμάτων. Πρέπει δηλαδή τα άνθρωπινα δικαιώματα να εγγραφούν στο επίκεντρο και τη προσέγγιση και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε αρκετές συνεδριάσεις προκειμένου. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε μέσα από την Επιτροπή μα ω προ τη Λιβύη. Αλλά όπω είπα ήταν κάποιε συνεδριάσεις στο θέμα ε, της ακτοφυλακή ε, αρκετά δύσκολες μια δεύτερη προσπάθεια μετά την, ε, την είδα που είχε προηγηθεί κάποιες εβδομάδες πριν. Ε, αυτά λοιπόν από τη Λιβύη. Όταν έρθει η ώρα θα τα ξαναπούμε. Έκθεση Νίγηρα. Τι θα λέγατε αντί να διαβάσω εγώ ε, μια μακροσκελή έκθεση ε, να ζητήσουμε από τους συναδέλφους που ήταν ε, στην αντιπροσωπεία για τον Νίγηρα. Και για να μην πλατιάζουμε, θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους είναι εδώ, ο Φρανκ ή ποιος άλλος. Μόνο εσύ, Φρανκ. Όχι μόνο εσύ δηλαδή. Είσαι τόσο σημαντικός, αλλά η Έρικα τα έχει φορτώσει όλα. Φαντάζομαι ότι συμφωνεί μαζί μου ο Φρανκ. Είχε και τη σχετική ευθύνη στην προετοιμασία μαζί με τη Λίδα και άλλους αυτής της ε, συνάντησης με βουλευτές από τον Αίγυρα. Όταν φτάσαμε το πρόγραμμα μας δεν ήταν τόσο δατικό όσο ήταν στο τέλος γιατί το προσαρμόσαμε για να το γεμίσουμε. Μπορέσαμε να συναντήσουμε. ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο ο κύριος Έγγελ αυτό. Συναντηθήκαμε με όσους θέλαμε να συναντηθούμε. Ήταν πολύ χρήσιμη η, η επισκέψη λοιπόν. Και παρακαλώ τον Φρανκ Έγγελ να λάβει το λόγο για να μας ε, ενημερώσει Για να προχωρήσουμε θα ζητήσουμε από τους βουλευτέ από τους προσκεκλημένου μας και όποιον άλλο ενδιαφέρεται. Το βελτιώσαμε στην πορεία και επικροτήκαμε σε λάθος σημείο γιατί αυτό κάνουμε στην, ε, στο Κοινοβούλιο. Γιατί ήταν η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, θέμα των αρχών ε, του Νίγηρα. Γιατί είναι χώρα διέλευση. Ε, μετανάστευση έχουν εδώ και αιώνε και θα συνεχίσουν να έχουν μετανάστευση. Και νομίζω ότι σε διάφορες συναντήσεις ε, υπογραμμίστηκε αυτό. Συναντήσεις οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί γύρω και μόνο, όπου το κράτος έχει αποτυχία. Υπάρχει ένα εδαφικό χάσμα, ένα εδαφικό κενό. Ε, και άλλες χώρες της περιοχής. Αυτό επαπειλεί λοιπόν όλους. Χαιρόμαστε λοιπόν που ο Νίγηρας ε, ακόμα αντέχει που ακόμα δεν δυνάμεις της για να μην καταρρεύσει όλος και να μην δημιουργηθεί ένα κενό εξουσίας. Γιατί οι κακές ειδήσει, ξέρετε, έχουν ε, περάσει μέσω της Βόρειας Αφρικής και εκεί. Η απειλή την υποστήριξή μας σε ό,τι αφορά την αντιστοιχή ε, η υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και έχω, έχω ε, επισκεφτεί και τη Μαυριτανία μια αλφα ασφάλεια στην επικράτειά του. Δεν το έχουν πετύχει αυτό στον Αίγυρα και στην Πουρκιναφθάσο και στο Βόρειο Τσάντ. Ε, έχουμε να το φροντίσουμε αυτό. Προσπαθούμε. Ευχαριστούμε Φράγκα, λέει ο Πρόεδρο. Έχουμε μια λεπτομερή έκθεση για τον Ήγηρα. Σα καλώ να τη διαβάσετε. Να επισημάνω κάποια σημεία κλειδί από πλευρά και τη αντιπροσωπεία σε σχέση με αυτά που είπε και ο Φρανκ και η Λίντα προηγουμένω. κατά την επίσκεψη στον Ήγηρα. Το βασικό θέμα που ανέκυψε είναι προφανώς η φτώχεια. Είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα του κόσμου ίσως. Το Μαλί έχει ξεσπάσει πόλεμος. Είναι πολλές οι χώρε που αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα. Άρα το θέμα για τον Νίγηρ από πλευρά μετανάστευση είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν φτάνουν καν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Νίγηρα είναι μια χώρα με τεράστια αντοχή παρά τι ε, πολλαπλέ προκλήσει τη φτώχεια και των άλλων ζητημάτων, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί χώρα διέλευσης. Δεν είναι μια χώρα που χρησιμοποιεί τους πολίτες της. Όταν περνάει ο κόσμος φυσικά από τον Νίγηρα, φυσικά και υπάρχουν πολλές επιστροφές, στρατατές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι σημαίνει το να είναι κανείς δίπλα στο θλιβί, τι σημαίνει να ζει κανείς δίπλα στο Τσάντ, ε, Μπουρκίνα Φάσο, Μποκοχαράμ, Λιβερία, με όλα τα προβλήματα που μαστίζουν τις χώρες αυτές. Και είδαμε λοιπόν ότι δείχνει το θέμα του πώς αντιμετωπίζει η Νίγηρα στα θέματα αυτά και τις βασικές υποδομές για την ανάπτυξη της χώρας. Δεν έχω, θεωρώ, συμμετέχει, συμμετάσχει ποτέ σε αποστολή με τόσο δεσμευμένους συνομιλητές και ομολόγους. Η σταθεροποίηση λοιπόν της ε, περιοχής είναι κρίσιμη. Συνδεθήκαμε και με την οικογόση. εξετάσαμε τι κάνουν και οι κορυφαίες πέντε χώρες στο Σαχέλ και με ΜΚΟ συνδεθήκαμε και την IOM, την υπατερμοστία του ΟΗΕ και πολλές άλλες ΜΚΟ, πάρα πολλές ΜΚΟ που εργάζονται επί τόπου και στην Ιγυρία και στην Αγκαντές. Διαβάστε παρακαλώ την έκθεση. Η ουσία όμως, το ζουμί είναι ότι πρόκειται για μια χώρα η οποία δεν εξαγάγει κόσμο, αλλά αποτελεί χώρα διέλευση από την, ε, την τη Λιβύη. Αντιμετωπίζει λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα και με χαρά θα ακούσω αυτά που έχουν να μας πούν και οι συνάδελφοι. Τα άλλα δύο μέλη της αντιπροσωπείας είναι η κυρία Κιέγγε και η κυρία Κοράτσα Μπίλτα. Αλλά δεν είναι εδώ στην αίθουσα, γι' αυτό λοιπόν θα, θα περάσουμε κατευθείαν στον πρέσβη, τον κύριο Ματέου Παουλά. Να σας ευχαριστήσω εκ νέου γιατί επί τόπου δεν ξέρω κατά πόσον συνάδελφοι έχετε συμμετάσχει σε τέτοιε αποστολέ, αλλά λίγο πολύ όλοι εξαφανίστηκαν όταν ε, μεταβήκαμε στη χώρα. Και εσείς φροντίσατε να συνδεθούμε με όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού. σα ευχαριστούμε λοιπόν, γιατί ξέρουμε ότι χάρη σε εσά σα στέφτηκε με επιτυχία αυτή η αποστολή. Σα ευχαριστώ πολύ και σε πέντε λεπτά αν θέλετε να μα κάνετε μια αξιολόγηση του που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, πρώτα πρώτα, ευχαριστώ γιατί οργανώσατε αυτή την αποστολή και επίσκεψη της ε, Επιτροπής σας στον ε, Νίγηρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την εταιρική μας σχέση, τη συνεργασία μας. Ευχαριστούμε επίσης για τη σημερινή πρόσκληση και έτσι διαπιστώνει κανεί πόσο δυναμικό χαρακτήρα έχει αποκτήσει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην με ακρηγορώ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι πολύ μεγάλα. Μερικά από αυτά ήδη αναφέρθηκαν, οπότε δεν χρειάζεται να με γρηγορήσω. Ασφάλεια και ανάπτυξη. Ε, Αυτά είναι τα κεφαλαιόδη ζητήματα, αυτά είναι οι λέξεις κλειδιά που αρχίζουν την κατάσταση στη χώρα. Ας ξεκινήσουμε με την ε, ανάπτυξη. Πρόκειται μάλλον για την πιο φτωχή χώρα του κόσμου. Ε, ανθεκτική, αλλά πάρα πολύ φτωχιά και επίσης ε, για να κάθε γυναίκα. Γι' αυτό που ανάπτυξη είναι πολύ προβληματικό. Για κατά προέκταση επιπτώσεις για το μέλλον της χώρας. Η τροφική ασφάλεια επίσης ειδικά βρίσκεται εν μέσω μιας πολύ ασταθούς περιοχής γιατί από τη μία έχουμε την ε, Λιβύη, από την άλλη έχουμε το Μαλί και την περιοχή της Μπόκο Χαράμ προς η χώρα, να υπάρχει κράτος και κρατικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια. Σε αυτά τα πλαίσια έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανταποκρίνει τα 690 εκατομμύρια ευρώ για το καταπίστευμα ε, για την περίοδο 14-20 υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ε, χέρι-χέρι με τις καταπίστευμα η ταμείο γιατί έχουμε και το θέμα της μετανάστευσης, έχουμε το θέμα του εμπορίου ναρκωτικών, να βοηθηθεί η κυβέρνηση να έχει περισσότερες δυνατότητες. Έχουμε επίσης και την αποστολή για το Σαχέλ και θα πρέπει χώρο ε, ε, αποστολές και κοινέ διοκτικές αρχές, ημών και ημών. Επίσης, τελευταία στο Νότο επιθέσεις του στρατιωτικού σκέλους της Μπόκο που ακόμη δεν έχει νικηθεί. Βεβαίως έχουμε κάνει τα να έχουμε επαγγελματική κατάρτιση κλπ. Τώρα όσον αφορά την μετανάστευση. Έχουμε το κατεπήγον ε, ταμείο, τους ε, δουλέμπορους, τους διακινητές ε, και όλη αυτή την παραοικονομία που έχει αναπτυχθεί για να βρουν κάποια δουλειά όλοι αυτοί οι Με λίγα λόγια, για να μην σε αυτά, είχα να σας ε, αναφέρω. Α, και η κατάσταση στη Λιβύα βεβαίως και μας έχει πλήρη παναπατρισμούς αυτού τις επιστροφές και για την ε, επανένταξη των μεταναστών όταν Ευχαριστώ και σας και την αντιπροσωπεία σας που ήρθε στη χώρα. Βόηθησε πολύ. Έτσι αναβαθμίστηκε. Έτσι θωρακίστηκε εταιρική μας σχέση με την Ευρώπη. Ε, και βέβαια και οι βουλευτές ε, που παρήσαν εδώ από τον Νίκη. Έχουμε την ε, αμήνα σε μήνους ε, δουλεμπορίας και το δίκτυο για την δημιουργία είναι τα δύο βασικά τα οποία μας απασχολούν. Αυτό με τη βοήθεια όλων των εμπλεκομένων για τη λάθρο μετανάστευση. Ξεκινώντας βέβαια από τους πιο νέους, η δεύτερη αποστολή. Και αυτό το άλλο είναι σημαντικό, να μπορέσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Έχει τρεις διαφορετικούς άξονες. Πρώτα, πρώτα, ανάπτυξη του δικτύου μετανάστευση. Παρά το ότι δεν έχουμε μετανάστευση προς την Ευρώπη. Λόγω της γεωγραφικής θέσης, ούτως ώστε να σταματήσει η λαθρομετανάστευση και να έχουμε αυτή την καταγεγραμμένη, την νόμιμη μετανάστευση. Και έμαθα τώρα ότι αυτή η συνάντηση πήγα στην Τίφα. Είναι μια περιοχή εκεί και με άλλες βουλευτίνες επισκεφτήκαμε αυτές τις γυναίκες. Πήγαμε στα στρατόπεδα προσφύγων. Θέλουν ε, να ζήσουν με ανθρωπιά, με ανθρωπιστικές συνθήκες. Πήγαμε σε τρία τέτοια στρατόπεδα καταβλισμού τέλο πάντων ένα εκ των οποίων έχει πάνω από 10.000. Ευχαριστούμε που το επισημάνατε. Ξέρουμε ότι πολλά θέματα σχετικά με τον υγεία δεν προχωρούν τις συνθήκες όπως ε, οι γυναίκες αυτές που είναι θύματα της Ποκοχάρα. Καλώς ήρθα τον ε, Μανού Αγκάλη, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Νίγηρα θεωρεί ότι έχει δύσκολη εκλογική περιφέρεια. Ο συνάδελφο έχει ω εκλογική περιφέρεια το Άγκαντα. ευχαριστούμε ιδιαίτερα λοιπόν που ήρθε και θα μα εξηγήσει τι συμβαίνει σε σχέση και με το, τη μετανάστευση και τους δρόμους του Αγκαντές. Έχετε το λόγο κύριε Σνάλφο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να έρθω να σας μιλήσω μετά την έκθεση για την κατάσταση στον Ήγηρα. Ευχαριστώ την ε, Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, τον ε, Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον Ήγηρα, όλους όσοι ήρθαν στον Ήγηρα, όλους όσοι είχαν την να μας υποδεχθούν εδώ. Θα αναφερθώ λοιπόν στον Ήγηρα, αλλά ξεκινώ από τη δεκαετία του 90 την αφήγησή μου. Ήταν η στιγμή κατά την οποία μία στάση έκλεισε με μια συμφωνία ειρηνευτική, με όρους καλούς, με όρους που τηρήθηκαν. Μία, ένας από τους όρους όμως συμφωνίας ειρήνης αυτής σήμαινε και την επανένταξη των ενόπλων. Αυτοί επέλεξαν μια ε, πιο, μια πιο επικερδή δραστηριότητα την ε, μεταφορά μεταναστών, υποψήφια μεταναστών. Εγώ τότε εργαζόμουν στην Υπατή Αρμοστία για την αποκατάσταση της ειρήνης. Είμαι από την περιοχή του Αγκαντές, ναι, αλλά έχω ασχοληθεί ειδικά με το θέμα αυτό της μετανάστασης σε μία περίοδο όπου έπρεπε σε αυτούς τους ένοπλους που είχαν ε, συνάψει την ενευτική συμφωνία να βρεθεί μια δραστηριότητα και βρήκαν τους μετανάστες, αυτούς που ήθελαν να έρθουν στην ε, Ευρώπη και, τους, ε, και ανέλαβαν να τους μεταφέρουν. Χωρίς αυτό να απασχολεί κανένα. Μια επόμενη στάση έφερε αντίστοιχα φαινόμενα και εξελίξεις. Και η κατάσταση δεν αλλάζει. Ο Νίγηρας δεν είναι χώρα προέλευσης, αλλά διέλευσης μεταναστών. Η πρωτεύουσα της ε, βόρειας χώρας, το Αγκαντές, έχει το νόημα της πόλης που και το ίδιο το όνομα Αγκαντές δηλαδή σημαίνει έλα να το επισκεφθείς και μετά ξαναφεύγεις αυτό σημαίνει η λέξη έτσι λοιπόν προχώρησε η ιστορία κατά τρόπον ώστε το 2015 έφτασε ο Νίγηρας να υιοθετήσει νόμο, το νόμο υπαριθμών 36, 036 του 2015, που καθιστά ποινικό αδίκημα την ε, δραστηριότητα μεταφοράς ή διευκόλυνσης της μετανάστευσης. Οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη μετανάστευση δηλαδή. Πρόκειται για ένα νόμο τον οποίο ε, έχει εισαγάγει η Δημοκρατία του Νίγηρα, χάρη στην ε, κυβέρνηση και τη διορατικότητα του Προέδρου μας, ε, Σουφού Μαμαλού, έχει εισαχθεί αυτή η νομοθεσία και τηρείται βέβαια στον ε, Νίγηρα, έχει ψηφιστεί και από την Εθνοσυνέλευση. Άλλο αντίστοιχο νόμος είναι ένας δίδυμος νόμος που έχει να κάνει με το εμπόριο ανθρώπων. Ε, είναι ακόμα βέβαια και τώρα πολλοί εκείνοι που θέλουν να πάρουν το δρόμο της μετανάστευσης και εκείνοι που είναι πρόθυμοι να τους βοηθήσουν. Αλλά αν κάνουμε μια, έναν απολογισμό της εφαρμογής του νόμου 036-2015 θα δούμε ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν γιατί ε, διέπραξαν αυτό το αδίκημα και έχουμε και ένα πρόγραμμα ε, Παναφορά στην νομιμότητα και αποκατάσταση ε, που αφορά αυτή τη στιγμή 5.655 συμπολίτε μα οι οποίοι θα αποδοθούν στην κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά έργα ε, υποστηρίξει για τα θέματα της μετανάστευσης, ε, της παράτυπης μετανάστευσης, για ευαισθητοποίηση, για ιδιαίτερη προστασία της παλαιάς πόλης του Αγκαδές, αλλά και για την εξασφάλιση όρων ε, κοινωνικής ενσωμάτωσης εκείνων που αναλάμβαναν την μεταφορά ε, και διακίνηση των μεταναστών. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν. Ε, υπάρχουν κυβερνητικέ οργανώσεις διεθνού εμβέλειας που δραστηριοποιούνται, Τις βλέπουμε, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευση, Οργάνωση Αναπτυξιακή Συνεργασία της Γερμανίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, Βεβαίω τα Ηνωμένα Έθνη με τις ε, υπηρεσίες τους μας βοηθούν όλοι αυτοί. ώστε να εξασφαλίσουμε την αναμετατροπή και απόδοση στην κοινωνία των πρωτεργατών αυτών ε, της ε, μετανάστευσης, παράτυπης μετανάστευσης. Εγώ έχω δηλώσει ότι εάν δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα της μετανάστευσης δεν έχει λόγο να ξανακλεκώ βουλευτής. Είναι κέριο ζήτημα για το Αγκαντές, για όλη μας την οικονομία, για ένα σύνολο πολιτών. Πρέπει να τους πείσουμε λοιπόν να αλλάξουν δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που βρίσκουν επικερδή γύρω από την οποία αναπτύσσεται μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων, γιατί ο ένας θα έχει το αυτοκίνητο, ο άλλος θα έχει το σπίτι, ο άλλος θα έχει το εστιατόριο, άλλος θα ετοιμάζει το πακέτο βασικού εξοπλισμού για το μετανάστη, θα έχει το ανταλλακτήριο συναλλάγματος. Μια, ένα ολόκληρο πλαίσιο λοιπόν δραστηριοτήτων και ήταν πολύ καλό το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργασία με την κυβέρνηση του Νίγηρα για την ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση αλλά και την εφαρμογή του νόμου για μας σήμερα είναι λόγος μεγάλης περηφάνειας η εφαρμογή αυτού του νόμου δεν 36-2015 όσοι είναι στο Αγκαδές έχουν, δεν έχουν πάει σχολείο το, το ξέρουν πολύ καλά το νόμο αυτό και είναι ένας τρόπος αυτός για να αντιμετωπίσουμε την παράτυπη μετανάστευση υπάρχουν επιτυχές και της ανάπτυξης οπωσδήποτε αλλά και όπως λέει άλλωστε και η έκθεσή σας, οι δραστηριότητες ε, που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια. Γιατί συμβαίνουν πολλά φοβερά πράγματα στην έρημο. Πεθαίνουν πολλοί γυναίκες, παιδιά εγκαταλείπονται. Η μετανάστες είναι αθώοι τελικά. Θύματα εκείνων που προσπαθούν να κερδίσουν στην πλάτη τους υποσχόμενοι ότι θα μπορέσουν να διασχίσουν την έρημο χωρίς κίνδυνο. Η έρημος είναι ένα τεράστιο νεκροταφείο όλων αυτών των υποψήφιων μεταναστών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, νέοι, μικροί, μεγάλοι, χρειάζονται τη δική μας υποστήριξη. Ναι, ναι, υπάρχει μετανάστευση, αλλά οργανωμένη, τακτή, ανθρώπινη, ε, με τρόπο οργανωμένο που θα έχουμε όλοι μαζί συμφωνήσει για να υπάρχει δυνατότητα για απασχόληση και μέλλον για αυτούς τους νέους. Έχω μιλήσει αρκετά, δεν ξέρω αν ο πρόεδρος μου επιτρέπει να συνεχίσω. Ας ολοκληρώσω εδώ. Ευχαριστώ και πάλι. Ήρθα να πω πολλά και να επαναλάβω ότι θα συνεχίσουμε τις επαφές. Πάνω απ' όλα όμως ήρθα να σας ακούσω και είναι μεγάλη για μας η περηφάνεια που είμαστε σήμερα εδώ ο Νίγηρας είναι χώρα διελεύσεως και όχι προελεύσεως. Και στέκουμε στα πόδια μας χάρη στους εταίρους μας και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως γιατί χάρη σε αυτούς στεκόμαστε ακόμα όρθιοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που και εσείς και εμείς που είσαστε εδώ σήμερα. Θέλαμε να κάνει λίγο παραπάνω ζέστη σήμερα στις Βρεξέλλες, αν και αυτό φαντάζομαι ότι δεν έχει σχέση με την ε, ζέστη που έχετε εκεί στη Σαχάρα. Τέλο πάντων, ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικά αυτά που μας λέτε και οι συνάδελφοι σίγουρα θα θέλουν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Και φυσικά ε, στην εγκατέσβαση έχουμε τον IOM και στην Τινιδά και στην ε, Λιβύη. Έχουμε πρόσφατα μεγάλη συμμετοχή του IOM και κ. Πατρίς Κασάντα είναι ειδικό σε θέματα ανταπόκρισης ε, από περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και θα μας ε, δώσει τη δική του ανάλυση. Για πέντε λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούμε ότι η επίσκεψη στο Αγκατές και στα κέντρα υποδοχής ήταν αρχά σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ της ε, εξέλιξης της αναπτυξιακής, ε, της ασφάλειας και της μετανάστευσης, συγγνώμη. Και με την προστασία της, με, την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων, κατέστη δυνατή αυτή η πρόοδος, με τα οποία ε, βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και κινδυνεύουν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης. Άρα ο αριθμός και βοήθειας για τα άτομα τα οποία έχουν ε, περάσει τέτοιες δύσκολες κατάστασεις σε προστασία, θέματα τρατότητας, υγεία. Μιλάμε επίσης για τις χώρες οικοβάς όπου υπάρχει η ηλεκτροκινητικότητα συσταγωγικά, σε ό,τι αφορά τα άτομα που θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους ε, σε πολύ... Έχασαν τη ζωή τους πρωτού φτάσουν οι αποστολές διάσωσης. Ξέρουμε λοιπόν τι χρειάζεται μα βοηθειά. Βλέπουμε ότι τι εννοούμε με την προστασία όταν δεν υπάρχει εναλλακτική μέσω νόμιμων οδών. Δύσκολο θέμα. Οι εξελίξεις ό,τι αφορά στην ασφάλεια. Οι συνάδελφοι μίλησαν ε, για την κατάσταση στον Ήγηρα και αντικείμενο διακινητών και βλέπουμε ότι κάποιες οικογένειες ήταν πιο εύκολο να πιστούν πρόσφατα, αλλά και υπάρχουν ε, και επιχειρήσεις οι οποίες θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι το θέμα της μετανάστευσης δεν θα συνδεθεί απόρριτα ναι. με το θέμα της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Ε. Είναι τα οποία τα είχαν πετάξει στην ερημό. Αν δεν τα είχατε λοιπόν βοηθήσει εσείς αυτά τα άτομα, πώς να σα το πω, δεν υπήρχε περίπτωση να κλειτώσεις την Άννα που είναι επικεφαλής των παγκόσμιων δράσεων και την καλωσορίζουμε. Αν θα θέλετε να πάρετε το λόγο και εσείς, Πάτρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πρόσκληση στην ε, συνάντηση αυτή και η παρουσία των συναδέλφων από την Ήγυρα. Είναι μεγάλη πρόκληση της μετανάστευσης και σίγουρα το αντιμετωπίσει το θέμα αυτό ο Νίγηρας, ε, το είπε και ο κ. Αγγελά άλλωστε. Έχουμε λοιπόν κάποια ενημερωτικά σημεία να σας ε, δώσουμε και να σας και μαζί σας κάποιες ανησυχίες που έχουμε. Όπως αναφέρθηκε η κατάσταση στον Ιγυραίο προφανώς συνδέεται με την κατάσταση στην Λιβύη και τον υπόλοιπο στις υπόλοιπες περιοχές. Πρόκειται για μια αναλλακτική ζώνη προστασίας για τα άτομα τα οποία έχουν διαφύγει από τη Λιβύη. Ξέρετε ότι γίνεται και ένωση σε πολλές περιπτώσεις στη Λιβύη. μετά από τις φρικτές συνθήκες κράτησης που επικρατούν στη Λιβύη. Ή άτομα τα οποία έρχονται από τη Λιβύη λόγω της πολύ δύσκολης κατάστασης στη Λιβύη ή άτομα τα οποία βρίσκονται στον Ήγηρα και σκοπεύουν να μείνουν. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να ανοίξω μια μικρή παρένθεση να σας πω ότι ο Νίγηρας αποτελεί μεν χώρα διέλευσης αλλά αποτελεί και χώρα ασύλιο, άρα και χώρα προορισμό, δυστυχώ. Για, 600, 60.000 υπηκός του Μαλή, ο Νίγρας αποτελεί χώρα ασύλου και για κάποιους έτοντες άσυλο και μετανάστες που δεν έχουν έρθει από τη Λιβύη αλλά έχουν ε, καταφτάσει κατευθείαν στον Ήγηρα και έχουν ζητήσει λοιπόν εκεί άσυλο. Ποιος είναι ο στόχος ε, και η στόχη α, του, της ύπατης αρμοστίας ε? να δοθεί μία αρρωγή και να βρεθούν ε, βιώσιμες λύσεις. Άρα ο Νίγηρας αναπτύσσει το σύστημα χορήγησης ασύλου κατά περίπτωση. Αλλά υπάρχει η σχετική νομοθεσία και υπάρχουν και τα θεσμικά όργανα προκειμένου να υπάρχει νόμιμη ε, καταχώρηση των ατόμων αυτών που καταφθάνουν και ζητούν άσυλο στη συνέχεια. Έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ο Νίγηρας ε, για κάποιες για ε, κάποια άτομα θέλουν να παραμείνουν στον ήγυρα. κάποια άλλα θέλουν να επαναγκατασταθούν εκτός της χώρας. Για παράδειγμα, για τα άτομα τα οποία έχουν εκενωθεί από τη Λιβύη, πάνω από χίλια άτομα έχουν εκενωθεί από τη Λιβύη, από την Τρίπολη προς την, τον ήγυρα με τη βοήθεια των αρχών του ήγυρα παρεμπιπτόντος. και ως τώρα 141 τέτοια άτομα έχουν ε, βρει μία λύση σύμφωνα με την ε, συμφωνία που έχει γίνει με το Νίγρα και περίπου 100 μετανάστες ε, έχουν εγκατασταθεί στον Νίγρα χωρίς να έχουν εκκληθεί από την Λιβύη. Το δεύτερο θέμα είναι το Αγκαντές, προφανώς το αναφέρεται και αυτό ένα σταυροδρόμι μετανάστευση ε, και η κατάσταση εδώ και κάποιου μήνες μας απασχολεί ιδιαίτερα. Περίπου 2.000 Σουδανοί βρίσκονται εκεί. Σουδανοί πρόσφυγε στη μεγάλη πλειοψηφία τους και ανελικοί ασυνόδευτοι και θύματα α, εκμετάλλευσης. Και πολύ φοβόμαστε ότι θα αυξηθούν δραματικά τα αριθμητικά αυτά στοιχεία τους επόμενους μήνες. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερως. Η Πατιαρμοστία έχει ανοίξει στο εγκατές λοιπόν γραφείο στα τέλη του 2017 και ένα οίκο αν θέλετε ένα σπίτι υποδοχής για τα πιο ευάλωτα άτομα. Όλα αυτά με τη συνεργασία της εθνικής, των εθνικών και περιφερειακών αρχών και όλους τους κοινωνικούς εταίρους και με την Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Τέσσερις είναι οι προκλήσεις τις οποίες διακρίνουμε στο άμεσο μέλλον σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Δεν μιλώ για τους ε, πρόσφυγες του Μαλή ή του Νιγηρά. Σε ό,τι αφορά την ε, Σουντανική ομάδα, όχι για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Κατά δεύτερον, όπως αναφέρθηκε επίσης, στο Κατές, αλλά και σε άλλα μέρα, ο ντόπιο πληθυσμός ε, προφανώς αισθάνεται ότι απειλείται από όλη αυτή την προσοχή που δίνεται στους πρόσφυγες. Μα της οικονομικής ε, ανάπτυξης, όπως αναφέρθηκε τρίτη πρόκληση. Τα άτομα τα οποία κοινωνούνται από τη Λιβύη, περίπου 8.000 στον αριθμό, αποτελούν αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή του Αγκαντές, έτσι ε, περαιτέρω. Ιδιαιτέρως γιατί μαζί με τις ε, αρχές της Βενησίας προκειμένου να μην ματρηθεί η αρχή της μη επιστροφής ε, σε ό,τι αφορά την επιστροφή δηλαδή ατόμων σε χώρες οι οποίες δεν είναι όμως ασφαλείς. Ευχαριστώ πολύ και είμαστε στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ε. Ευχαριστώ. Τέλος να ακούσουμε και τους δύο εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ε, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλές εθνικές και τοπικές ΜΚΟ αλλά να ακούσουμε καταρχάς ε, τον κύριο Χαβό από τον Ερυθρό Σταυρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά του να μην κανείς τελευταίος. Βέβαια, μια που ακούσαμε τόσο πλήρω. Τι να πω να σας τα πω γαλλικά, πάντως σημειώσουμε στα αγγλικά είναι. Και όπως ξέρουν οι συνάδελφοι από την Νιγηρία, ο ο Ερυθρός Σταυρός έχει μια στιβαρή παρουσία στη χώρα και έχουμε εννέα φορείς ε, προχη τροφίμων, ασφάλεια, επομένως διατροφική, αλλά και βοηθούμε τις οικογένειες ε, γενικότερα στα πλαίσια των μας, οπότε είναι η δραστηριότητά μας ε, αρκετά έντονη και επίσης πλησιώνουμε τους μετανάστες ε, όσον αφορά τα υγειονομικά, την ε, κοινωνική πρόνοια, επίσης ε, τους μαθαίνουμε τα βασικά των πρώτων βοηθειών και εδώ και χρόνια επίσης έχουμε δραστηριοποιηθεί στα Εκεί υπάρχει βεβαίω πολλή πορνεία και επομένως έχουμε αναπτύξει δραστηριότητα όσον αφορά σχετικές ε, δοκιμές για οροθετικούς ε, κλπ. Με τη βοήθεια του Δανέζικου Ρεθροσταυρού ε, σε επίπεδο επεμβάσεων ιατρικών. Τώρα πέραν της Επιτροπής θα πρέπει να πούμε για τους αδέλφους ότι είχαμε με τον IOM ε, ανταλλαγή θεμάτων πρέπει να διεκπαιρεώσει ο ένας και ο άλλος φορέας. Επίσης έχουμε και το Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό στην χώρα και φροντίζει για την επανένωση οικογενειών και γενικά την πλαισίωση όλοι εκεί να προσαρμοστούμε στις τοπικές άνοιγες όπως άλλωστε ισχύει παντού και έχουμε έτσι κάποιες κινητές μονάδες γιατί βέβαια διστάσουν μετανάστες να πάνε στα κέντρα υγείας. Οπότε με τις κινητές μονάδες πλησιώνουμε να λάβετε υπόψη λίγο το ότι ε, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, επεκτείνει κάποια προγράμματα. Αλλά έτσι τις άμεσες ανθρωπιστικές ανάγκες όπως αυτές που εμείς παρέχουμε όπως είπαμε για υγεία, υγιεινή και θα πρέπει να βοηθήσουμε βέβαια. Κάθαρο ότι έχει μειωθεί σημαντικά η ροή μεταναστών. Η εφαρμογή του νόμου 2015 έχει προφανώς συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ροής μεταναστών μέσω των ήγερα προς τη Λιβύη και την Ευρώπη. Ξέρετε κύριε και κύριοι βουλευτές, ως ανθρωπιστική οργάνωση θέλουμε να πούμε ότι η εφαρμογή του νόμου και τη ευεργετική αριθμητικά τουλάχιστον. Δηλαδή οδήγησε στην ε, μείωση των τακτικών ροών μεταναστών. Έχει παρόλα αυτά συνέπειες για τους ανθρώπους τους ίδιους και θέλουμε να σας ενημερώσουμε είναι όλο και πιο κατασταλτικό καταρχάς το κλίμα κατά των μεταναστών και πιο επιθετική η πιο έντονη η βία που χρησιμοποιεί η αστυνομία εις βάρος των μεταναστών στο δρόμο της μετανάστες. Αυτό βλέπουμε και από όσα μας λένε οι μετανάστες και από, τα, συζητήσεις μαζί τους δηλαδή το διαπιστώνουμε γιατί μας λένε ότι προπυλακίζονται, δέχονται ε, ταπεινώσεις, βασανιστήρια, τραυματισμούς ακόμη. Επίσης, ο νόμος αυτός έχει μετατρέψει τον μετανάστη σε λαθρεπιβάτη του Αγκαντές. Επομένως, οθείται προς τα περίχωρα του Αγκαντές, αλλά και προς την, ε, τα άκρα της ε, περίθελψης, δηλαδή ούτε σε ιατροφαρμακευτική φροντίδα έχει πλέον, ακόμα και σε φαγητό δεν έχει σχεδόν πια πρόσβαση, γιατί φοβάται να βγει να φάει, μην τυχόν και τον συλλάβουν. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρόβλημα της μεταφοράς των μεταναστών και της εξώθησής τους ε, στο περιθώριο των ε, κοινωνικών παροχών. Γιατί βλέπουμε και το είπαμε ότι είναι όλο και λιγότερο μετανάστες, αλλά και αυτοί που υπάρχουν, ε, εάν αρρωστήσουν μέσα στον κέτο και τους πούμε πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο να σας φροντίσουν, φοβούνται, φοβούνται να πάνε. Μόνο όταν είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση πάνε σε κάποια μονάδα υγειονομικής περιθέρψης κρατική. Επιπλέον και όλο και περισσότερο ενδύνονται οι κίνδυνοι για τους μετανάστες. Πολύ είναι πολύ πιο υψηλοί από ό,τι στο παρελθόν. Όποιοι λαθροδιακινητές, δηλαδή τολμούν ακόμη να διακινήσουν μετανάστε, ε, ζητούν πιο πολλά χρήματα. Η επιβίωση των μεταναστών τους εγκαταλείπουν στην έρημο. Αρκεί να μπορέσουν να ξεφύγουν από τη δίωξη από την αστυνομία. Μια εικόνα που τελικά επιδεινώνει την κατάσταση για τους μετανάστες, συνθήκες διαβίωσής τους στην πόλη του Αγκαντές. Ελπίζουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, Κέστερ, Στέτινα, Σπινέλη, Λάμπερτ, καλά όλοι δηλαδή. Παρακαλώ, ε, ξέρω βέβαια ότι με μεγάλη υπομονή κάτσατε και παρακολουθείτε, αλλά όσο το δυνατόν σύντομα. Πάνω απ' όλα θέλουμε να δώσουμε χρόνο στους ε, βουλευτές που ήρθαν από τόσο μακριά να απαντήσουν στις παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Η Επιτροπή λοιπόν παρακαλώ και μετά ο κύριο Πέστερ ε, πρώτος. Τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσκληση να μιλήσουμε. Νομίζω ότι η πλήρης παρουσίαση της κατάστασης ε, συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση προόδου στην εφαρμογή της ατζέντα για το έγγραφο αυτό παρουσιάζει λοιπόν μια συνεκτική προσέγγιση στη μετανάστευση σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο, σε ό,τι αφορά και το διεθνές δίκαιο και σε συνεργασία με τους ε, συναδέλφους από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και από την υπατηρμοστία του ΟΗΕ όθηση του συστήματος υποδοχής ε, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Όλες αυτές οι προσπάθειες λοιπόν γίνονται παράλληλα. Η επιλογή να συμπεριληφθεί και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θεωρώ ότι αποτέλεσε μια σωστή επιλογή για το άτομα τα οποία επανακαταστάθηκαν και από τα κράτη, τα δικά τους κράτη να σας μιλήσω για το μέλλον στη Λιβύη και τον Ήγηρα. Στη Λιβύη το θέμα είναι να συνεχιστεί το πρόγραμμα επανεκατάστασης. με κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για το μηχανισμό επίγουσας διέλευσης. σε ό,τι αφορά την πολιτική δέσμευση από την Αφρικανική Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ομάδα Εργασία του ΟΗΕ, η ύπατη άρμοστη δραστηριοποιείται στην Τρίπολη για να διευκολύνει την εκένωση από τη Λιβύη. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε λοιπόν οικονομικά την ε, προσπάθεια αυτή και τα κέντρα υποδοχής ε, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για να υπάρξουν στον Ήγηρα. Να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε για το κοινοβουλευτικό δίκτυο για τους μετανάστες και για την ιστορία της νομοθεσίας του ΣΠΑΙΡΑ για να δοθούν οικονομικές, ε, οικονομική υποστήριξη και υποστήριξη σε ό,τι αφορά τις θέσεις απασχόλησης. Έχω μαζί με την Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ε, προωθούμε την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της βίας. Έχουμε ως τώρα πάνω από 500 δικαιούχους που έχουν καταρτιστεί σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης. Είναι λοιπόν αυτή μια απτή έκφραση των όσων έχουμε συζητήσει και όσων ζητήσατε προηγουμένως υποστήριξη της οικονομίας και υποστήριξη της χώρας. Δεν θα, αναφέρω στο, δεν θα αναφερθώ στο καταπίστευμα γιατί ήδη αναφέρθηκε και δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, επιβεβαιώσουμε ότι ο Νίγηρας ε, έχει πάρει στα σοβαρά αυτή την πρωτοβουλία για τη βελτίωση της συνεργασίας των χώρων στην περιοχή σε θέματα ασφάλεια και μετανάστευσης και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργάζεστε και για την μείωση των ροών των μεταναστών που περνούν από τη χώρα, αλλά και την εισρωή. Πρόεδρε, μου ζητήσατε να είμαι σύντομη και μια και κάποια στοιχεία ήδη αναφέρθηκαν από του ε, άλλου ε, συναδέλφου, Θα κλείσω στο σημείο αυτό. Εμεί ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, να μίλησατε για τη δουλειά σας, αλλά Ε, μου έλεγε και η κυρία Μακαμένα ότι έχουμε συναδέλφους από την ε, ΕΚΟ και άλλες υπηρεσίες οπότε μπορούν να μας συμπληρώσουν την ε, εικόνα αλλά να δώσουμε λόγο τώρα στον κύριο Κώστα Κύριοι εμπειρογνώμονες, κύριοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου του Νίγηρα, λέει ο κύριος Κώστερ, σήμερα ακούσαμε τόσα πολλά για το οποίο σας ευχαριστούμε και ο προηγούμενος είναι θετικός, δηλαδή ότι τον τελευταίο χρόνο για το Σαχέλ ενδιαφέρει και έκανε πολλά η Ένωση και τα κράτη-μέλη. Όμως το θέμα είναι ότι ίσως δεν είναι βιώσιμες αυτές οι λύσεις γιατί πολλές φορές δεν βοηθούμε τις χώρες Αφρικής να βρουν τις λύσεις μόνες τους. Ε, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να μεταθέτουμε στις χώρες αυτές την Ευρώπη φρούριο για να κρατήσουμε μακριά τους μετανάστες. Οπότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες τελευταία ε, έχουν ως κίνητο των ενεργειών τους το φόβο εναντί του μεταναστευτικού. Προσπαθούν να βρουν ε, λύσεις εντός εισαγωγικών, ούτως ώστε να φρενάρουν τους Αφρικανούς από τη μετανάστευση. Και πολλές φορές τέτοιες πολιτικές οδηγούν σε ανθρωπιστικές τραγωδίες. Άρα τελικά καταλήγουμε να έχουμε λένε και περισσότερους μετανάστες οι οποίοι αφήνουν πνοή στη διαδρομή όπως μας είπατε. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι η πολιτική και η οικονομική αστάθεια νοτίως της ε, Σαχάρας είναι άμεσο αποτέλεσμα της ε, απικιακής εκμετάλλευσης, της επικιοκρατίας. Ε, Είτε δηλαδή η ιδιοποίηση των φυσικών πόρων οδήγησε σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Με τίποτα δεν έχουμε πιο ανθρωπιστική στάση. Και για τον Ήγερα και για άλλους χώρους στην περιοχή. Η λύση δεν είναι εξοπλισμός. Όχι να κουκουλώνουμε τους νεκρούς. Έχουμε αυτή την πολιτική ασφάλεια εντό εισαγωγικών, οπότε δεν αφήνουμε την ελευθερή διακίνηση στην περιοχή του ΕΚΟΒΑΣ ακόμα και αν ε, εκεί είναι μια ελεύθερη περιοχή, δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσε και ε, ο συνάδελφος ή συνάδελφοι από τη χώρα μας τα εξηγήσουν. Γιατί έτσι έχουμε περισσότερη αστάθεια. Έτσι έχουμε ριζοσπαστικοποίηση. Δεν είναι δυνατόν να πετύχουμε την ασφάλεια και την σταθερότητα μόνο με βοήθεια ε, στο στρατό. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι προοπτική για τους νέους νοτίους της Σαχάρας. Και επίσης να αναγνωρίσουμε ότι είναι γείτονε, ότι είναι εταίροι μας μετά από τόσα... Κύριε Κιώστερ, πολύ καλά τα είπατε, πρέπει λίγα λεπτά για να μπορέσουν να μας τα πούν ξανά ευθύς που των ακούσαν οι προσκεκλημένοι μας. Έχετε το λόγο. Πάρα πολύ σωστό είναι να ακούμε την αλήθεια για το τι συμβαίνει εκεί επί τόπου. Είναι συγκλονιστικό να ακούμε σε τι συνθήκες κινούνται εκεί οι μετανάστες και αυτοί που τους πλησιώνουν είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι γίνεται στην πράξη. Είναι σταθερή η χώρη σας. Δεν θέλει να φύγει ο κόσμος λέτε. Μπράβο σας. Αυτό σημαίνει ότι έχει επιτελέσει σημαντικό έργο. Οπότε πάλι μπράβο γιατί βοηθάτε τι γίνεται με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλείνεται με τις εντάσεις που δημιουργούνται μεταξύ μεταναστών και ντόπιων. Και ξέρετε, έχω σπουδάσει στην ανθρωπολογία και έχω διαπιστώσει στους καταβλισμού μεταναστών εδώ στην αξίωσή τους γιατί είναι πάρα πολλοί οι νέοι που ήρθαν και με βρήκανε για να μου πούν για τους ε, μήνες, τα χρόνια που πέρασαν για να φτάσουν στην Ευρώπη. Όλοι μίλησαν επίση για τις business που έχουν αναπτυχθεί περί το μεταναστευτικό όλους ε, δικού σα πόσο έχει ε, τελικά καλύψει αυτούς που έρχονται. Αν μπορείτε, πέστε μας για αυτό το διαβόητο νόμο του 10 που ποινικοποιεί τα πάντα τα σχετικά με την μετανάστευση. Κυρία Σπινέλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Η Ευρώπη θα πρέπει να τηρήσει τα υποσχεθέντα. Πρώτα πρώτα το θέμα της μετεγκατάστασης αυτών των ε, ναι, για... και τελικά οι μετακαταστάτες ήταν μόνο 30. Στην αρχή του Μαρτίου τους σε μου είναι ότι αυτή η στρατιωτική βοήθεια είναι δυσάλογα μεγάλη οι επιπτώσεις όσον αφορά επίσης την ρύθμιση των ροών, τη δράση των λαθροδιακίνητων που απασχολούν τον Ερθρό Σταυρό και τους γιατρούς του κόσμου. Κύριε Σαρτζεντίνη. Α, Λάμπερτς πρώτα. Κατόπιν κύριε Σαρχεντίνη. Παρακαλώ ένα δύο λεπτά για να μπορούσαμε να έχουμε χρόνο οι προσκεκλημένοι μας να μας ε, μιλήσουν. όπως ξέρετε, έχουμε και άλλη ακρόαση μετά. Σας ευχαριστώ. Έχω ένα-δύο θέματα που επαφές ε, και τη συνεργασία, τοπική κοινότητα και κοινωνική συνοχή είναι το θέμα μου. Ε, για την ε, βία από την αστυνομία. Βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά